Good morning everybody. We will start. Καλημέρα σε όλους. Comenzamos la, la reunión de hoy. Θα αρχίσουμε με τη σημερινή μας συνεδρίαση. Το θέμα 9, σημείο 9, ανακοινώσει της Προέδρου. Ε, μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση των συντονιστών ε, με διάφορα σχόλια και θέσεις που εκφράστηκαν. Κατανομή η ε, εξέσεων ιδίες πρωτοβουλίας Οι συντονιστές της ομάδας σας έχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες και ποιοι θα είναι οι εισηγητές και θα μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες αυτές σε εσά. Και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το 10. Πρόκειται για την έκθεση περί ισότητας άντρων γυναικών το 2013 με εισηγητή τον κύριο Ταραμπέλα. Του δίνουμε το λόγο αμέσως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, αναφέρθηκε και κατά τη διάρκεια της πρώτης ανταλλαγής απόψεων. Θέλω αυτή η έκθεση να είναι αποτελεσματική και διαρθρωμένη σε τέσσερα θέματα. Ε, Ευρωπαϊκή Ένωση 2020, οικονομική διάσταση, ο ρόλος γυναίκα γυναίκας στην κοινωνία είναι ο πρώτος άξονας. Θα εστιάσουμε στην απασχόληση των γυναικών και στην φτώχεια, την επισφάλεια ορισμένων γυναικών, συνταξιούχων κλπ. Δεύτερον, συμβασμός ε, μεταξύ ιδιωτικής και, δημοσιακής και επαγγελματικής ζωής. Τρίτον, η βία κατά των γυναικών. Και τέταρτον, τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την στρατηγική Ευρώπη 2020, ε, έχουμε στόχους για, τη, για μια οικονομία ε, βιώσιμη ευφύ και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να πάρουμε μέτρα υπέρ της απασχόλησης των γυναικών. Στόχος ήταν 75% το 2020, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 63% απασχόληση γυναικών, μακριά από το στόχο μας. Στην προηγούμενη έκθεση, έκθεσή μου, το 2010, πριν από 5 χρόνια, ε, ε, η απασχόληση ήταν 59,1%. Δηλαδή έχει αυξηθεί λίγο, παρόλο τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Τώρα πρέπει να δούμε και την ποιότητα της απασχόλησης βέβαια. Θα πρέπει να πάρουμε μέτρα υπέρ, μιας, υπέρ ποιοτικών θέσεων εργασία, μείωση ε, την διαφορών στους μισθούς, ε, διαφάνεια στους μισθούς, καταπολέμηση ε, των στερεοτύπων ε, και αποφυγή εμποδίων στην εξέλιξη των γυναικών τόσο σε ό,τι αφορά την άνοδό τους όσο και την διεύρυνση των τομέων στους οποίους προσλαμβάνονται δηλαδή οριζοντίως και κατακορύφως. Τρίτον, να δούμε ποιες είναι οι, οι ανάγκες τους, ε, οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν λάβει ε, εκπαίδευση ποιότητας ή που αρνούνται να ε, μετεκπαιδευτούν, να επιμορφωθούν κλπ. και δυσκολεύονται να βρουν θέση εργασίας μετά. Δεύτερος άξονας, η φτώχεια. Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να μειώσει κατά 20 εκατομμύρια τα άτομα τα οποία πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό εξοπλισμό. Στις μονογονεϊκές οικογένειες το 91% αυτών είναι η γυναίκα αυτή που αναλαμβάνει τα παιδιά και όπως και οι συνταξιούχες και αυτές οι γυναίκες μονογονεϊκών οικογενειών ε, ζουν σε μια επισφάλεια πιο αυξημένη σε σχέση με τους ε, άντρες. ε, μία στις τέσσερις γυναίκες ζουν σε επισφάλεια, ένας στους έξι άντρες. Ε, η φτώχεια των παιδιών οφείλεται στην επισφάλεια των γονιών τους πολύ συχνά. Για να πετύχουμε το στόχο της μείωσης φτώχειας θα πρέπει να μειώσουμε τις διαφορές μεταξύ των συντάξεων που αυτή τη στιγμή φτάνουν στο 39% ε, πιο μεγάλη διαφορά μεταξύ των συντάξεων από τη διαφορά μεταξύ των μισθών. Ε, πολλές γυναίκες ε, ηλικιωμένες δεν έχουν καν σύνταξη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αλλάξουν επίσης το φορολογικό τους σύστημα για να λάβουν υπόψη την εξέλιξη της δομής των οικογενειών. Έτσι ώστε οι μονογενικές οικογένειες και οι ηλικιωμένοι να μην τιμωρούνται. Θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν στρατηγικές ένταξης πιο ισχυρές. Τρίτον, συμβασμό μεταξύ της ιδιωτικής και της επαγγελματικής ζωής. Ε, ε, συμφιλίωση. Ε, για τις γυναίκες φαίνεται να είναι πιο δύσκολη η συμφιλίωση, αλλά και οι άντρες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ε, πάντως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συμφιλίωση αυτή ε, και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Η Κομισιόν και τα κρατημέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα όπως να ξεπεράσουν τους στόχους της Βαρκελόνης για να προσφέρουν οι υπηρεσίες φύλαξης παιδιών ε, με οικονομικό τρόπο αλλά και ελαστικά ωράρια εργασίας. Δεύτερο μέτρο, ε, πατρική άδεια. Εφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προσφέρουν τέτοιου είδου δυνατότητα, άδειας για τον πατέρα δηλαδή όταν γεννιέται ένα παιδί. Η, Ελλάδα και το Λουξεμβούργο προστείνουν μόνο δύο μέρες την άλλη μεριά. Ε, και βέβαια εκείνη την εποχή που γεννιέται ένα παιδί αρχίζουν ε, τα ζευγάρια και μοιράζονται τους ρόλους. Επίσης ζητούμε τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν περισσότερο ε, τη θέση του πατέρα σε ό,τι αφορά τις γονικές άδειες. Χρειάζονται νομικά και, ε, και μη νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα λοιπόν για να μπορέσουν και οι πατεράδες να συμφιλιώσουν την ιδιωτική τους ζωή με την επαγγελματική τους ζωή. Αυτό θα βοηθούσε και τις μητέρες. Ε, η άδεια μητρότητας από την άλλη μεριά είναι και αυτή ένα ζήτημα τόσο ό,τι αφορά τη συμφιλίωση της ιδιωτικής με την επαγγελματική ζωή όσο και την απασχόληση. Ε, μια μητρική άδεια επιτρέψει οι γυναίκες να κάνουν παιδιά και μετά να επιστρέψουν στην επαγγελματική του ζωή. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συνεργαστεί με το Συμβούλιο γιατί τα κράτη-μέλη ασφαλώς ε, δεν έχουν ε, μετακινηθεί σε σχέση με τις παλαιότερες θέσεις τους, δεν έχουν κάνει και πολλά πράγματα αλλά και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει πράγματα. Ε, πιστεύω δηλαδή ότι και εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια συνένεση εδώ, εντό, εδώ εντός του Κοινοβούλου για να πιέσουμε αποτελεσματικά και το Συμβούλιο. Ε, το θέμα αυτό βρίσκεται σε στασιμότητα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το ξεμπλοκάρουμε και εδώ εντός του Κοινοβουλίου και στη συνεργασία μας με το Συμβούλιο. Τρίτο, τρίτος άξονας, βία κατά των γυναικών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ε, της Υπηρεσίας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, μία στις τρεις γυναίκες ε, στην Ευρώπη έχει υποστεί ε, σεξουαλική ή άλλου τύπου βία. Το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να πιέζει την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη έτσι ώστε πρώτον να επικυρώσουν την σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη το σύντομο το δυνατό. Αυτή τη στιγμή μόνο 8 χώρε τον κάνει: η Δανία, Αυστρία, Γαλλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία. Και οι υπόλοιπε χώρε πρέπει να κάνουν το ίδιο. Και βέβαια μετά θα πρέπει να την εφαρμόσουν κιόλας αυτή τη σύμβαση. Δεν αρκεί απλή, απλώς η υπογραφή, η επικύρωση. Δεύτερον, ε, να εγκαθαρίσουμε μια Ευρωπαϊκή Μέρα για τη βία κατά των γυναικών. Ε, το πρότεινα για το το, το, το πρότεινα και παλαιότερα, ε, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή της κοινή νόμης σε ένα θέμα το οποίο πολύ συναντεύεται στα φώτα της δημοσιότητας. Και δεύτερον θα μας επιτρέψει ένα τέτοιο έτος ε, να υποφεληθούμε των βέλτιστων πρακτικών. Τρίτον, να συλλέξουμε συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα, στατιστικά. Και τέλος, μια οδηγία πλαίσιο για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. Τέλος, αναπορικά και σεξουαλικά δικαιώματα. Είναι σημαντικό το ζήτημα. Ε, θα πρέπει η θέση μας να επαναβεβαιωθεί. Το κείμενο το οποίο έχω αναφέρει είναι ακριβώ το ίδιο με αυτό που υιοθετήσαμε στην προηγούμενη μου έκθεση το 2010, στις 10 Φεβρουαρίου του 2010. Εκεί υπήρχε ένα, μια παράγραφος που ε, αναφερόταν στο δικαίωμα των γυναικών ε, να χειρίζονται όπως επιθυμούν το σώμα τους και να έχουν πρόσβαση σε αμβλώσεις και αντισύλληψη. Ε, αυτή η παράγραφος είχε γίνει δεκτή, ε, δεκτή με 368 ψήφους υπέρ και 237 ψήφους κατά. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα το παρόν κοινοβούλιο είναι πιο προοδευτικό από το προηγούμενο, οπότε φαντάζομαι ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Ε, Παρ' όλα αυτά η έκθεση δεν είναι πλήρης, διότι θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σε σχέση με το θέμα μας, ε, να μην παρεκκλίνουμε, ε, αλλά μπορούμε να προσθέσουμε και κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, για την ιδιαίτερη θέση των γυναικών γεωργών των αγροτησών. Ε, δεύτερον, ε, η αχειραφέτηση των γυναικών δια, της, δια του του αθλητισμού. Τρίτον, γυναίκες και έρευνα. Ε, όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσω τροπολογιών. Ε, περιμένω τις προτάσεις σας. Θα ήθελα να καταλήξουμε σε μια ισορροπία όμως. Το κείμενο προφανώς είναι ανοιχτό, ε, μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις, αλλά παρακαλώ πολύ αποφύγεται, να αποφύγουμε αυτό το κείμενο να γίνει χριστουγεννιάτικο δέντρο όπου μπορούμε να κρεμάσουμε οτιδήποτε, οποιοδήποτε στολίδι. Ε, οπότε στις τροπολογίες σας παρακαλώ πολύ να σεβαστείτε τη δομή της έκθεσης και να είστε όσο πιο ε, συνοπτικοί και συνοπτικές και αποτελεσματικοί γίνεται. Ε, στην... Ε, προηγούμενη θητεία μας ε, πολύ συχνά πλήταμε την εικόνα μας ε, γιατί μέσα σε εκθέσεις μας βάζαμε πολλά πράγματα τα οποία λεπικαλύπτοντο, δεν είχαν άμεση σχέση με το θέμα κλπ. Το 2014, στην αρχή του 2014, ε, ε, ε, δεν έγινε δεκτή η έκθεση για την ε, σχέση μεταξύ, ε, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν ήταν καλό το, το αποτέλεσμα αυτό. Οπότε ας προσέξουμε αυτή τη φορά. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 9η Δεκεμβρίου σε μία εβδομάδα. Δεν ξέρω αν είναι μεσημέρι ή μεσάνυχτα. Οπότε ε, παρακαλώ μέχρι την 8η Δεκεμβρίου να έχετε στείλει τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ταραμπέλα. Στα αρχικά έγγραφα, σε, στην, στην πρώτη εκδοχή των εγγράφων δεν μπορούμε να βάλουμε όλα τα πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας. Ε, υπάρχει περιορισμός, οπότε μπορεί μετά να εμπλουτιστεί το κείμενο μέσω της συζήτησης. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα καταρχήν για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Ταραμπέλα για τη δουλειά του εδώ και πολλά χρόνια υπέρ της ισότητας των φίλων. Να τον ευχαριστήσω για το, την πλήρη αυτή έκθεση που μας υποβάλλει και την οποία μας παρουσίασε. Δεν πρόκειται να επαναλάβω θέματα τα οποία ανέφερε. Θα εστιαστώ σε ορισμένες από τις ε, τροπολογίες που θα υποβάλω. Συμφωνώ γενικά με την έκθεση, θέλω απλώς να τη συμπληρώσω. Η καλύτερη κατάρτιση των γυναικών δεν σημαίνει βελτίωση της απασχόλησης και βελτίωση ποιότητας ε, των θέσεων εργασία των γυναικών. Ε, ξέρουμε πώς είναι αυτοί που έχουν πανεπιστημιακά πτυχία ε, το 60% αυτών είναι γυναίκες, δεν το βλέπουμε αυτό στην απασχόλησή τους, ούτε στους μισθούς τους, ούτε στην ποιότητα των θέσεων που προσφέρονται στις γυναίκες. Συνεπώς, υπάρχει ένα διαρθρωτικό θέμα. Ε, θα πρέπει να δούμε λίγο τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε επίσης σε ό,τι αφορά θέματα όπως διαφήμιση. Οποιαδήποτε εφημερίδα και αν πάρετε σήμερα ε, στην Ευρώπη Κοιτάξτε τι, διαβάστε τι οπουδήποτε, οποιαδήποτε εφημερίδα στην Ευρώπη. Ε, οι, οι πρώτες, οι βασικές ειδήσει ε, έχουν σχέση με άντρες. Παρόλο ότι υπάρχουν και γυναίκες ε, που εργάζονται στην πολιτική κλπ, οι γυναίκες πάντοτε είναι δεύτερες ειδήσει ή κοινωνικές ειδήσει. Πρέπει να Βελτιώσουμε επίσης λέμε τις, τους μισθούς και τις, ε, τη, τις θέσεις απασχόλησης αλλά δεν θα πρέπει να αγνοούμε, να παραμελούμε και τα καθημερινά. Ε, συνεπώς η διαφήμιση, η γλώσσα που χρησιμοποιούμε ε, είναι σημαντικά ζητήματα. Ε, η επιστημονική κατάρτιση είναι πολύ σημαντικό θέμα επίσης. Χρειαζόμαστε ε, ιδιαίτερες πολιτικές έτσι ώστε οι γυναίκες να επιλέγουν ε, επιστημονικές ε, εξειδικεύσεις. Εμείς στη χώρα των Βάσκων τι έχουμε κάνει. Έχουμε προσπαθήσει να φέρουμε σε επαφή τις γυναίκες με τον επιστημονικό κόσμο έτσι ώστε οι γυναίκες να εμπνέονται και να επιλέγουν τέτοιου τύπου σχολές. Γιατί αυτές στην πράξη οι σχολές δίνουν τις πιο ποιοτικέ θέσεις εργασία. Συνεπώς, επιστημονική κατάρτιση, επιστημονική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Μετά, υπηρεσίες για τις γυναίκες έτσι ώστε να συμφιλειώσουν την ιδιωτική με την επαγγελματική ζωή. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη φροντίδα των ηλικιωμένων, γιατί όλες οι εκθέσεις ευρωπαϊκό επίπεδο λένε ότι οι γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για το, τη φροντίδα των ηλικιωμένων από ότι άντρε. Συνεπώ ναι, τη φροντίδα των παιδιών, αλλά μην ξεχνάμε και τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Μετά, συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια θα πρέπει μια, μια ακόμα φορά να επιδιώξουμε και την πολιτική συμμετοχή με ίσους όρους. Συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό, ασφαλώς, παντού και στην τέχνη, στη μουσική κλπ. Υπάρχουν παντού διακρίσεις ε, και μην ξεχνάμε να κάνουμε μια αναφορά και στις γυναίκες με αναπηρίες, οι οποίες ε, πλήττονται από μια διπλή ανισότητα. Συμφωνώ επίσης με όσα ελέγχθησαν για τη βία. Το θέμα όμως είναι διαρθρωτικό. Οι εκθέσεις λένε συνεχώς ότι μια καλύτερη εκπαίδευση των ατόμων ε, δεν θα οδηγήσει σε κατάργηση της βίας. Υπάρχουν ε, ε γυναίκες που είναι θύματα ανθρώπων ε, που προέρχονται από οποιαδήποτε κοινωνική τάξη και μορφωτικό επίπεδο. Συνεπώς θα πρέπει να το δούμε ως διαρθρωτικό πρόβλημα και αυτό. Οπότε γενικά είμαστε υπέρ της έκθεσης, θα πρέπει όμως να εναρμονιστεί η νομοθεσία περισσότητας μεταξύ άνδρων και γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί υπάρχουν ακόμα ευρωπαϊκές χώρες που θεωρούν ότι τα θέματα της ισότητας και το θέμα της ε, βίας ε, κατά των γυναικών είναι θέμα ιδιωτικού δικαίου και όχι δημοσίου δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε μια εναρμόνιση της νομοθεσίας περισσότερα των δύο φύλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές ήταν οι τροπολογίε μου. Ευχαριστώ πολύ ξανά τον κύριο Ταραμπέλα με βρίσκει πολύ σύμφωνη η έκθεσή του. Muchas gracias, señora Bilbao. Les eh, pido a partir de este momento que intenten hacer intervenciones eh, reducidas en el tiempo porque todavía nos quedan tres puntos eh, que tratar en el orden del día antes eh, del comienzo de, de la comisión. De... Παρακαλώ πολύ να είστε πιο σύντομοι γιατί μας μένουν ακόμα τρία θέματα ε, και έχουμε μετά τη κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Madame la, la Présidente. Euh, je vais m'exprimer au nom de notre euh, rapporteur fictif. Ε, παίρνω το λόγο εκ μέρους της σκιώδης ηγέτρας της Μαρίας Γκαμπριέλ. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ταραμπέλα για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Θεωρεί ότι η έκθεση του κ. Ταραμπέλα πραγματικά σχολιάζει και περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά θέματα. Θέμα για παράδειγμα της ίσης αμοιβής ανδρών γυναικών ε, στο πλαίσιο 2006, ε, η καταπολέμηση των στερεοτύπων των σχετικών με το φύλλο, η σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας. Το θέμα της ε, ανάγκης καταπολέμησης όλων των τύπων βίας κατά των γυναικών, ε, επικύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, ανάγκη ε, συμφωνία στο Συμβούλιο για το θέμα της συμμετοχής των γυναικών στο, στα διοικητικά συμβούλια κλπ. Όλα αυτά τα θέματα ο κ. Σταραμπέλα τα ενέταξε πολύ σωστά στην έκθεσή του Η έκθεση αυτή είναι πραγματικά πολύ ισορροπημένη και πετυχαίνει τους στόχους που έχουμε θέσει. Η κυρία Γκαμπριέλ θα ήθελε να προτείνει και κάποιες τροπολογίες για να ενισχύσουμε ε, ορισμένα σημεία της έκθεσης. Καταρχήν σε ό,τι αφορά την ε, διαφοροποίηση ε, ε, των τύπων καριέρας που ακολουθούν οι γυναίκες. Ε, δεύτερον, ε, στην καταπολέμηση των ε, στερεοτύπων και στην, ρόλο της εκπαίδευσης σε αυτήν. Τρίτον, συγκεκριμένα μέτρα που χρειάζονται για την βελτίωση της συμφιλίωσης μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματική ζωής. Έτσι και αλλιώς ο κύριος Ταραμπέλα αναφέρει ότι αυτή η συμφιλίωση αφορά εξίσου τους άντρες και τις γυναίκες. Συνοψίζοντας, αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι η ακτές είναι πολύ ισορροπή. Η σκιώση γήτρια του Έλκη, κυρία Γκαμπριέλ, ε, εκφράζει μια ευχή, μια επιθυμία. Οι συνάλφοι να ε, είναι προσεκτική σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των τροπολογιών που θα ε, προτείνουν όπως ζήτησε και ο κύριος Ταραμπέλα έτσι ώστε η έκθεση αυτή να μην γίνει χριστουγεννιάτικο δέντρο όπως είπε ο εισηγητής. Ε, θα πρέπει να προτείνουμε τροπολογίες με νυφαλιότητα, ε, να είμαστε λυτοί, προσεκτικοί έτσι ώστε να αποφύγουμε το, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν πέρσι. Ε, να αποφύγουμε δηλαδή ή, να υποσκάψουμε το έργο μας. Εμείς, ε, η κυρία Γκαμπριέλ μάλλον, ε, θα είναι πολύ επικοδομητική και θα συνεργαστεί με τον κύριο Ταραμπέλα έτσι ώστε η έκθεση να υιοθετηθεί και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια και να οδηγεί σε μια βελτίωση της ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, προς την κατεύθυνση της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λεγκρίπ. Κυρία Νταντσέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ταραμπέλα για την εξαιρετική του εργασία και για την διάρθρωση όλων των σημείων που πρόβαλε, αλλά και για το ότι περιέλευε και πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω ορισμένες πτυχές. Καταρχάς, τη διάκριση κατά των γυναικών ε, είναι αποτέλεσμα και των αντιλήψεων που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Υπάρχει μια μεγάλη ανισορροπία στην αγορά εργασίας η οποία πολλές φορές καταλήγει σε διακρίσεις και έχει επιπτώσεις στο θύμα των διακρίσεων, στον αποδέκτη των διακρίσεων. Πραγματικά θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία σαφή αντίληψη δεδομένου ότι υπάρχει σαφώς, υπάρχουν σαφώς φως μεγάλης διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων. Πολλές φορές οι γυναίκες πρέπει δεν έχουν την εμπειρία των ανδρών οι οποίοι πολλές φορές φεύγουν και εργάζονται μακριά από την οικογένεια ενώ οι γυναίκες πολλές φορές είναι πιο πολύ στο σπίτι ε, και δουλεύουν, ε, έχουν οικιακές απασχολήσεις ε, κλπ. Συμφωνώ με τον εισηγητή ε, και με αυτά που είπε ότι θα πρέπει να έχουμε μια έκθεση που να περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές επιτυχίες, τα πιο σημαντικά προβλήματα χωρίς να είναι υπερφορτωμένη η έκθεση και θα πρέπει να αντανακλά μια ισόρροπη και ουδέτερη ε, περιγραφή των, της καταστάσεως. Eh, Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τους συναδέλφους και με την άποψή τους ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να είναι πιο ισόρροπη. Ο κύριος Ταραμπέλε είπε ότι δεν μπορεί να συμπεριλάβει τα πάντα και όλα αυτά τα οποία είχε προγραμματίσει. Δέχομαι και χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρόταση του να ξαναρχίσουν οι διαβουλεύσεις για την οδηγία ε, της ε, γονικής ε, άδειας. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και στην Ήπεθρο, στις γυναίκες που απασχολούνται στην Ήπεθρο. και σε αγροτικές περιφέρειες όπως και η, η απλήρωτη οικιακή εργασία. Ξέρουμε ότι πολλές φορές γυναίκες, μητέρες με οικογένεια ε, δουλεύουν ατελείωτες ώρες ε, στο σπίτι σε οικιακή απασχόληση που δεν αναγνωρίζεται πουθενά. Θα πρέπει λοιπόν να αναφερθεί αυτή η απλήρωτη οικιακή εργασία και να προτείνουμε οι γυναίκες να μπορούν να γυρίσουν πίσω στις εργασίες τους μετά από τη μητρική άδεια. Δυστυχώς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό το δικαίωμα ε, ε, επανένταξης στην εργασία δεν δίνεται και οι γυναίκες αποκλείονται. Στο σημείο 14 αναφέρει ο κύριος Ταραμπέλα ότι αυτό το σημείο είναι αντίθετο με τα δικαιώματα των κρατών μελών. Ε, είναι όμως γεγονός ότι οι αμβλώσεις δεν αποτελούν θέμα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητος. Το δικαίωμα στη ζωή είναι επίσης και ένα δικαίωμα ε, ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Επίσης, δεν αναφέρει αυτή η έκθεση τις μεγάλες διαφορές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας ανδρών και γενικό παραδείγματο χάρη την έγκαιρη ε, προ... Ε, ε, επισήμαση και πρόληψη του καρκίνου πολλές φορές θα, πρέπει να δίνεται η ευκαιρία και άδεια στις, ε, στους εργαζόμενους ε, να πηγαίνουν για μια εξέταση κατά τη διάρκεια της εβδομάδος ε, ιατρική εξέταση δηλαδή. Πο, πολλές φορές δεν έχουν τον καιρό να, να προσφύγουν σε, σε έναν γιατρό να γίνει μια απαραίτητη εξέταση διότι απασχολούνται στη δουλειά και στο σπίτι. Πιστεύω λοιπόν τελικά θα καταλήξετε, λαμβάνοντας υπόψη παρατηρήσεις, σε μια καλή, καλύτερη έκθεση. Η κυρία, ο κύριος Μπάστιαν. Καταρχήν, να ζητώ συγγνώμη, συγγνώμη ε, ε, γιατί ο κύριος ε, ε, δεν είναι παρόν. Ε, μιλώ εγώ εκ μέρους της ομάδας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ταραμπέλα Ιδίω σε ό,τι αφορά την δομή του εγγράφου που το καθιστά πολύ κατανοητό. Χαιρόμαστε που συμπεριλήφθησαν τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα και ιδιαίτερως που ζητούμε να ξεμπλοκαριστεί η ε, οδηγία για τις γυναίκες σε ε, ψηλές ε, δικτικές θέσεις και η οδηγία για την μητρότητα. Ε, επίσης χαιρόμαστε που ε, οθούνται οι, ε, παροτρύνονται χώρες που δεν το έχουν κάνει να υπογράψουν τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Θέλουμε να υπογραμμιστούν κάποια θέματα χωρίς να αμφισβητούμε την δομή και την ουσία της έκθεσης. Θέλαμε να υπογραμμιστεί περισσότερο το θέμα των συνεπειών των γυναικών, επί των γυναικών, των περικοπών στο, στα συστήματα στα κοινωνικά συστήματα και γενικότερα της ε, ε πολιτικής λιτότητας. Εγώ προέρχομαι από την ε, Ισπανία που έχει ακολουθήσει μια τέτοια πολιτική ε, λιτότητας ε, και έχουν πληγεί ιδιαίτερα γυναίκες. Επίσης θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 να συμπεριλάβει έναν απολογισμό ε, της, ε, της ισότητας ε, των μέτρων που έχουν ληφθεί έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε συγκεκριμένες συστάσεις για το μέλλον. Επίσης το θέμα του φύλου θα πρέπει να συμπεριληφθεί και σε άλλες, σε άλλες διαδικασίες όπως τα μία Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τέλος, είναι σημαντικό να δούμε την να δούμε από πιο κοντά το θέμα της διαφοράς των συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό έχει σχέση με τη φτώχεια. Εν πάση περιπτώσει χαιρόμαστε που έχει συμπεριληφθεί ε, το θέμα της δημοσιονομικής πολιτικής και το πώς επηρεάζει την ισότητα των δύο ε, θα πρέπει επίσης να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο θέμα της διαφοράς, των διαφορών προκύπτων στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να ζητήσει τέλος την ε, Κομισιόν να ε, προτείνει ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο για τον, τον αγώνα κατά της βίας εναντίον των γυναικών. Επίση, παρόλο ότι είναι περίπλοκο, θα προσπαθήσουμε να είμαστε και εμεί ε, συνοπτικοί και σύντομοι στι τροπολογίε που θα υποβάλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην κυρία Χέιτ. Ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε ήδη πολλά πράγματα. Θέλω όμω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Ταραμπέλα για το πολύ καλό έγγραφο. Βέβαια πολλά θα μπορούσε και θα ήθελε κανεί να συμπεριλάβει ακόμα, αλλά η δομή του εγγράφου είναι πολύ καλή και τονίζω ότι είναι σημαντικό να μην αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα όπως την προηγούμενη θητεία προκειμένου περί αυτών των προβλημάτων. Εμείς στην Επιτροπή μας πρέπει να ταχθούμε υπέρ της ισοτιμίας ανδρών και ισότητας ανδρών και γυναικών, να προβάλλουμε τα δικαιώματα των γυναικών ε, και τα δικαιώματα πάνω στο σώμα της. Ε, νομίζω ότι θα υιοθετηθεί στην Ολομέλεια η εκθεσία αυτή. Ευχαριστώ. Για να τελειώσουμε την συζήτηση θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Ταραμπέλα. Παρακαλώ να είναι σύντομος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μπιλμπάου Μαραντίκα και όλους τους υπόλοιπους που συμμετείχαν και υπέβαλαν τις προτάσεις τους. Ε, από την κυρία Πετήρ ε, συγκράτησα διάφορες ε, ενδιαφέρουσες ιδέες, για παράδειγμα την πρόληψη. Δεν συμφωνούμε πάντοτε με την κυρία Πετήρα, αλλά είμαστε και δύο μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και εκεί σίγουρα ε, βρίσκουμε πολλά κοινά σημεία. Ε, πιστεύω ότι όλες οι προτάσεις ήταν επικοδομητικές. Ε, θα προσπαθήσω, ε, αφού πάρω τις τροπολογίες, ε, να τροποποιήσω το κείμενό μου έτσι ώστε πραγματικά να γίνει δεκτό από μια ευρεία πλειοψηφία. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρή Ραπό, την Μαραμό, την βοηθό μου, προς την οποία αν θέλετε μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με ε, αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι ήμουν σύντομος, Πρόεδρε. Όχι, κύριε Ταραμπέλα, δεν παραπονιέμαι. Έχουμε 10 ακόμα λεπτά. Ο κ. Ταραμπέλα το είχε αναφέρει, εν πάση περιπτώσει το επαναλαμβάνω και εγώ, την προθεσμία... Ε, για τις τροπολογίες αυτές είναι η 10 ε, Δεκεμβρίου. Ε, αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. Ε, ας δούμε αν μπορούμε να τελειώσουμε αυτή τη συζήτηση σύντομα. Υπεύθυνη κυρία Κούνεβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αντίλωτη εργασία πλήττει κυρίως τις γυναίκες όσον αφορά τη δουλειά στο σπίτι και σε μεγαλύτερου ανθρώπου. Χτε κατά τη συνεδρίαση τη Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων, άκουσα με προσοχή την παρουσίαση των εισηγητή τη σχετική έκθεση κ. Πύρισκη, ο οποίο υιοθετεί μια πολύ καλή προσέγγιση στο κείμενό του είναι σημαντικό πώς θέλει να πάμε ένα βήμα παραπέρα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να μην περιορίσουμε δηλαδή στην καταγραφή και πρόληψη του προβλήματος, αλλά να συμβάλλουμε ώστε να μετατρέψουμε την αντίλωτη εργασία σε νόμιμη εργασία. Οι προτάσεις που πιστεύω πώς μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία της πλατφόρμας είναι οι εξής. Η πρώτη τροπολογία αποδεικνύει ότι ακριβώς επειδή οι γυναίκες θίγονται πολύ περισσότερο από την αντίλωτη εργασία των όταν δουλεύουν στο σπίτι, όταν φροντίζουν ηλικιωμένους και παιδιά, χρειάζεται να γίνει πολύ προσεκτική καταγραφή αυτού του πληθυσμού κάθε χώρας και των μέτρων που θα πρέπει να λάβει κάθε κράτος μέλος για να αντιμετωπίσει αυτού του είδους την αντίλωτη εργασία. Με τις τροπολογίες 2, 3, 5 και 9 προτείνεται να έχει ρόλο να συμμετέχει και να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων. Η πλατφόρμα που θέλουμε να δημιουργήσουμε θα πρέπει μεταξύ άλλων να βοηθάει τους εργαζόμενους να ενταχθούν στο κοινωνικό πλαίσιο των αγορών εργασίας. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλά συχνά προβλήματα όταν διεκδικούν τυπικές θέσεις εργασίας. Έτσι αναγκάζονται να δεχτούν θέσεις αντίλωτης και επισφαλής εργασίας και να, επιβιών, και να επιβιώσουν και μπορούν να μεγαλώσουν έστω και με περιορισμένα μέσα τα παιδιά τους. Η συμμετοχή του Ινστιτούτου στην πλατφόρμα διασφαλίζει πώς θα λαμβάνεται υπόψη και οι ειδικέ πτυχές το φαινόμενο της αντίδοτης εργασίας όταν αφορά τις γυναίκες. Με την τοπογεία 4 εισάγουμε στις θεματικές ομάδες εργασίας της πλατφόρμας τα ειδικά ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες Παράδειγμα, όπως είπαμε και πιο πριν, μελέτη της παροχής οικιακών υπηρεσιών, η φροντίδα παιδιών και των ηλικιωμένων. Η εργασία αυτή συχνά δεν ελέγχεται, έχει επιπτώσεις στη κοινωνική ασφάλιση των γενικών. Η τροπολογία 6 είναι η σημαντικότερη. Προτείνει την υιοθέτηση από την πλατφόρμα ενός σαφούς ορισμού για την αδίλωτη εργασία. Ο ορισμός βάσει το οποίο δουλεύουμε χρονολογείται από το 1998. Αν θέλουμε η πλατφόρμα να είναι αποτελεσματική και χρήσιμη, θα πρέπει ο ορισμός αυτός να επαναξιολογηθεί. Χρειαζόμαστε όταν έναν ορισμό που περιγράφει πληρέστερα το φαινόμενο και μπορεί να ακολουθεί την εξέλιξη των παρατυπίων. Πιο συγκεκριμένα σήμερα και ακριβώς λόγω των κυρώσεων που επιβάλλουν κάποια κράτη-μέλη αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο της μερικής αντίλωτης εργασίας. Δηλαδή κάποιοι εργοδότες δηλώνουν μεν τους εργαζόμενους τους, αλλά όχι όλες τις ώρες εργασίας, ούτε για την πραγματική απασχόλησή τους. Αυτά όχι μόνο διονύζει τα προβλήματα που θέλουμε να, να αποφύγουμε, αλλά έχει και σαν αποτέλεσμα την βελτίωση των εθνικών δικτών με τρόπο πλασματικό. Με τις τροπολογίες 7, 8, 10, Υπενθυμίζουμε πως το φύλλο πρέπει να συμπεριληφθεί κατά την αξιολόγηση του φαινομένου της αντίλωτης εργασίας. Στην πραγματικότητα, η αγορά εργασία στι χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαχωρισμένες με βάση το φύλλο. Γυναίκε απασχολούνται συχνά σε τέτοιες εργασία που δεν είναι μόνο αντιλωτέ αλλά και μικρότερης διάρκειας, με λιγότερες ώρες εργασίας και με ελάχιστη αμοιβή. Αυτό δεν επιτρέπει σε αυτές τις γυναίκες να είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Λίγα στοιχεία είναι ωστόσο διαθέσιμα για να υποστηριχτούν πολιτικές που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Υπάρχει δε και έλλειψη στοιχείων σχετικά με την θέση των γενικών μεταναστών. Αν θέλουμε να ενισχυθεί η απασχόληση και να διασφαλιστούν τα εργασικά και κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών, πρέπει πρώτα να διασφαλίζουμε πώς μπορούν να εργαστούν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κούνεβα. Θεωρούμε ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση για αυτή την έκθεση. Ε, φτάνουν σιγά σιγά οι συνάλφοι της Επιτροπής ε, ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Οι τροπολογίες πρέπει να καταδεθούν μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου και σε αυτή την περίπτωση. Και αν ολοκληρώσουμε την κοινή μας συνεδρίαση με την Τροπή ΛΥΜΠΕ νωρίτερα από ό,τι έχει προβλεφθεί, μπορούμε να συνεχίσουμε με τη συζήτηση, καθώς και με τα άλλα δύο θέματα, σε ό,τι αφορά την απαλλαγή του προπολογισμού του 2013 ε, αν ολοκληρώσουμε νωρίτερα τη συζήτησή μας θα συνεχίσουμε αυτά τα θέματα. Αλλιώς ε, οι τροπολογίες και για, όλα τα θέματα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Οκ, okay, διακόπτουμε για μερικά λεπτά λοιπόν.